Good, good morning. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Επί συνάδελφη Αρχή συνεδρίαση με έξι λεπτά καθυστέρηση έχω να πω. Σας καλωσορίζω όλους θερμότατα. Ε, αυτή αίθουσα είναι από τις μεγαλύτερες που διαθέτουμε. Και 9 η ώρα σας πέφτει λίγο πρωί από ό,τι βλέπω. Τουλάχιστον οι καμπίνες είναι γεμάτες. Καλωσορίζω τους διερμηνείς που μας χαιρετάνε από μακριά και από ψηλά. Εδώ κάτω είναι αραιές οι γραμμές. Παρ' όλα αυτά οι σημαντικότεροι συνάδελφοι είναι παρόντες, δηλαδή δύο συνεισηγητές, μέχρι και αντιπρόεδρο έχουμε παρούσα και μερικούς συντονίστας. Καλωσορίσατε θερμά. Χαιρόμαστε που σήμερα έχουμε την ευκαιρία να συνεδριάζουμε για δεύτερη φορά. Ε, παρουσία του Προέδρου, συγγνώμη, Επιτρόπου κυρίου Μοσκοβισή, που είναι αρμόδιος και για τη φορολογία μεταξύ άλλων, τα τελευταία δύο χρόνια και στην Ολομέλεια αλλά και στις ειδικές εξεταστικές επιτροπές τάξη 1 και 2 και στη δική μας συζητούμε την τρέχουσα φορολογική πολιτική. Στις 14 Μαρτίου σε μια συζήτηση στην Ολομέλεια παρουσιάσατε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουν περάσει έκτοτε 7 εβδομάδες και στο μεταξύ μεσολάβησαν πολλές συνεδριάσεις για μεμονωμένα θέματα και σήμερα έχουμε στη μερίσια διάταξη μια φορά θέματα, μια σειρά από θέματα μάλλον ε, ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα. Για όλους εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα για να μπορούμε να διαμορφώσουμε ίδια άποψη. Τα έγγραφα που μας έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτιώνονται όλο και περισσότερο, φίλο, να ομολογήσω. Τα έγγραφα τα οποία είναι προσβάσιμα μόνο μετά από συνένεση του ε, Συμβουλίου χειροτερεύουν συνεχώς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το briefing note, το ενημερωτικό σημείωμα, της 20ης Ιουλίου 2016 για τον κώδικα δεοντολογίας. Ένα έγγραφο λοιπόν το οποίο δημοσιεύθηκε ή μάλλον κατατέθηκε αφού είχαν ολοκλώσει εργασίες τους οι επιτροπές Ταξ 1 ε, και 2. Είναι 33 σελίδων και με εξαίρεση την πρώτη σελίδα και την ημερήσια διάταξη όλες οι υπόλοιπες είναι μαύρες. <laughs> Γιατί θεώρησαν ε, ότι είναι το θέμα εσωτερικό, δεν αφορά το κοινοβούλιο, το οποίο αποδηγετούμε εμείς και χειραγωγούμε. Είναι ε, ένα έγγραφο εσωτερικό της ομάδας εργασίας και δεν επιθυμούμε να το δημοσιεύσουμε. Και λέω ειλικρινά, ε, τράξα μια φωτογραφία από μια μαύρη σελίδα, μαυρισμένη, γιατί αν καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, είναι μόνο μαύρο, τίποτα άλλο. Ε, το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να δέχεται τέτοια πράγματα, κύριε Επίτροπε. Δεν μιλώ για εσά, αλλά για το Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε τέτοιε καταστάσεις. Και είμαι απόλυτα αποφασισμένος να μην το δέχομαι έτσι σε αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με τα δικά σα έγγραφα που έχουν διαβιβαστεί και είναι και μεγάλη διαδικασία και βαριά να τη διαβάσει κανεί αυτή ε, τη βιβλιογραφία. Τα άλλα έγγραφα είναι κατάμαυρα. Σας έδειξα εδώ ένα ακραίο παράδειγμα. Λοιπόν, επανέρχομαι στις ερωτήσεις τις οποίες σας στείλαμε. Και εσείς ε, μας απευθύνετε μια απαντητική επιστολή. Και πριν κάνω και άλλα ε, προκαταρτικά σχόλια, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να μας κάνετε μια εισαγωγή και μετά να συζητήσουμε. Σας καλωσορίζω και πάλι. Παρακαλώ, έχετε μέσα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Βέρνερ Λάγκεν. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Δέχομαι τις προσκλήσεις σας πάντα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και έρχεται σε πολύ καλή στιγμή. Είναι πραγματικά σωστός ο χρόνος για να συναντηθούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την φοροδιαφυγή, τον, τον κοινό μας στόχο μετά από την ακρόαση του Δεκεμβρίου. Έχω λοιπόν την πεποίθηση ότι η μάχη στην οποία έχουμε εμπλακεί, τα δύο μας θεσμικά όργανα είναι φυσική σύμμαχη και σε σχέση με το πολιτικό κομμάτι, είναι σύμμαχοι φυσικοί και στα πλαίσια της αντίληψης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στα πλαίσια της αναζήτησης της διαφάνειας. Σε ό,τι λοιπόν περνάει από το χέρι μας, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής είναι η απόλυτη προτεραιότητα θα έλεγα ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει αυτό εδώ και δυόμιση χρόνια που συνεργαζόμαστε Το θέμα αυτό το έχουμε εξετάσει με φιλόδοξο τρόπο και μέσω επίσης της συνεργασίας με την δική σας Επιτροπή και με την προηγούμενη, την ΤΑΞ, εγώ τη συνεργασία αυτή προσπάθησα να την καταστήσω υποδειγματική αν αυτό είναι δυνατόν. Οι Ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να μας στέλνουν το μήνυμα απαιτητικό για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Το θέμα δεν είναι η επικαιρότητα μόνο. Τα Panama Papers βέβαια στον χρόνο σιγά σιγά χάνονται. Αλλά δεν θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο σκάνδαλο για να αντιδράσουμε οργανωμένα. Ας συνεχίσουμε με συστηματικό και έμμονο θα έλεγα τρόπο την εργασία μας. Νομίζω ότι αυτό θέλει το κοινοβούλιο σας. Θέλουμε να κατανοήσουμε ότι η πλειοψηφία των πολιτών της Ένωσης θέλει να δώσουμε τη μάχη α, της φοροδιαφυγής. Αυτό μας το ζητούν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το 74% των Ευρωπαίων πολιτών. Λοιπόν, σε προκαταρτικά να σταθώ σε τέσσερα θέματα. Πρώτον, πλησιάζει η στιγμή όπου θα αρχίσουμε να συλλέγουμε τους καρπούς της πρωτοβουλίας μας εξορισμού υπάρχει πάντα ένας νεκρός χρόνος. Από τη στιγμή που ξεκινά μια πρωτοβουλία νομοθετική, από τη στιγμή που η πρωτοβουλία αυτή μετατρέπεται σε ψηφοφορία και ψήφισμα και από τη στιγμή που εφαρμόζεται. Το 2017 λοιπόν θα είναι μια χρονιά για συγκεκριμένες δράσεις καρά της φοροδιαφυγής. Το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συλλεγεί πληροφορίες για τους λογαριασμούς και από το τέλος του 17 και μετά θα υπάρχει αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων. Δεν είμαστε μόνοι, 108 χώρες το κάνουν αυτό μετά από αποφάσεις που έχουν ληφθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτοί που κρύβουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό κάποια στιγμή θα αποκαλυφθούν. Όπως το είπα και στη Βέρνη την προηγούμενη εβδομάδα και στον Ελβετό Υπουργό, το τραπεζικό απόρριτο κάποιοι θα το νοσταλγήσουν ίσως, αλλά είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά εξαφανίζεται. Νομίζω ότι είναι ένα βασικό στοιχείο και μια βασική κατάκτηση για την οποία θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Όπως επίσης και οι εκθέσεις αναχώρα, όπως επίσης και οι αναφορές για τις ειδικέ φορολογικές ρυθμίσεις οδηγούν ε, στις ε, σωστές ανταλλαγές πληροφοριών δεν θα είναι εύκολο, αλλά νομίζω ήδη από το 2017 θα έχουμε μια πρώτη εφαρμογή όλου αυτού του πλαισίου. Νέες νομικές ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στις φορολογικές αρχές να χρησιμοποιήσουν στοιχεία για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος. Όλα αυτά θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2017. Νομίζω ότι αυτά τα οποία είπα σχεδιάζουν, ε, μορφοποιούν ένα νέο τοπίο νομοθετικό και πολιτικό. Βρισκόμαστε στην φάση κατά την οποία η εφαρμογή των προτάσεών μας, το implementation, θα πρέπει να προχωρήσει. Δεν θα πρέπει να μείνουμε σε αυτά τα οποία έχουμε κάνει ήδη και η πρωτοβουλία αυτή όπως και η νομοθετική πρωτοβουλία δεν θα πρέπει να αποτύχουν. Και ε, σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να διευρύνουμε και την εμβέλεια των δράσεών μας, χωρίς να χάσουμε βέβαια τον πυρήνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ελέγξει τη σωστή εφαρμογή και μεταφορά της οδηγίας, αλλά οι εσδήποτε δικητικές πρακτικές αντίθετες με το πνεύμα ε, της πρότασης δεν μπορούν να ανοιχνευθούν παρά μόνο μέσω ενός ε, κατάλληλου λογιστικού ελέγχου ή μιας καταγγελίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να προκαλέσει τέτοιου είδους ενέργειες. Είναι λοιπόν κεφαλαιόδες για την αποτελεσματικότητα της δράσης μας. Οι διαδικασίες οι μεταβατικές να ολοκληρωθούν με σωστό τρόπο. Είναι σημαντικό λοιπόν και είναι ρόλος δικό σας και της Επιτροπής να ασκηθεί πολιτική πίεση επί των κρατών μελών έτσι ώστε να συλλέξουμε τον καρπό της νομοθετικής μας πρωτοβουλίας. Δεύτερον, έχουμε τρεις προτεραιότητες καθορισμένες για τον υπόλοιπο του 17 και χρειαζόμαστε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι δεν σας κρύβω. Ο κατεπήγων χαρακτήρας των σκανδάλων τα οποία έχουμε περιγράψει, μερικές φορές με το χρόνο χάνεται το ενδιαφέρον για αυτά. Καταρχάς, το CCCTB με τη νέα του μορφή πρόκειται για ένα διαφθρωτικό σχέδιο με μια διπλή διάσταση, μια διάσταση που αφορά στην εσωτερική αγορά, στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στη διαφάνεια κατά καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αν συνδυάσουμε το CCCTB με την οδηγία αυτή, αυτό θα απαγορεύσει στις επιχειρήσεις να μεταφέρουν τα κέρδη τους προς τους φορολογικούς παραδείσους. Λοιπόν, έχουμε ανάγκη από το CCCTB και στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Παρά τις ανακοινώσεις τις οποίες έχουμε κάνει μέχρι τώρα και παρά τις συναντήσεις τις οποίες κάναμε εδώ και ένα περίπου χρόνο, και τη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μνούτσιν των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Σύμβουλο επί των Οικονομικών του Ντόναλτ Τραμπ, τον κύριο Γκάρικον, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις, ε, απορίες θα έλεγα καλύτερα, για τους προσανατολισμούς της νέας Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει με προληπτικό τρόπο να προωθήσει την διεθνή ε, οικονομική διακυβέρνηση. Ε, στις δύο συναντήσεις της ομάδας των 20 είχαμε αρκετά προβλήματα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν αποχωρήσει από την πολυμερή διάσταση, θα ήταν ψέμα. Δεν έχουν στραφεί στον αυστηρό προστατευτισμό, θα ήταν επίσης ψέμα και το ίδιο ισχύει και για την απόσυρση των Αμερικανών από τις συνέπειες της, τη μάχη για τις συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών. Πάντως τα πράγματα αλλάζουν σε σχέση με τη μορφή των παραδοσιακών τρόπων συνεργασίας δεν υπάρχουν αντιστάσεις, αλλά από την άλλη δεν διαπιστώνουμε και μια κάποια ιδιαίτερη δυναμική και ενθουσιασμό. Υπολογίζω λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργαστούμε σωστά και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στον τομέα του CCTB το ταχύτερο δυνατόν. Δεν θα πρέπει να χάσουμε την όθηση την οποία έχουμε. Να το πω αλλιώς, αν δεν βοηθήσετε τα πράγματα θα είναι δύσκολα γιατί υπάρχουν επιφυλάξεις, κάποιες από αυτές ε, τις κατανοώ, κάποιες άλλες τις εξηγώ αλλά δεν τις υιοθετώ. Η τρίτη προτεραιότητα είναι ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Φορολογικών Παραδείσων. Εδώ θα πρέπει να στοχεύσουμε στο σωστό επίπεδο φιλοδοξίας. Γνωρίζω ότι για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας μέχρι το τέλος του 2017 θα πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος των λεγόμενων μη συνεργαζομένων φορολογικών δικαιοδοσιών έτσι ώστε να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει τα κράτη-μέλη έτσι ώστε η λίστα αυτή να συνταχθεί μέσα στις σωστές προθεσμίες. Τώρα, Πρέπει να πούμε πόσο σημαντικό είναι το μέσο αυτό στα πλαίσια της διεθνούς εμπλοκής μας για την χρηστή ε, διεθνή διακυβέρνηση. Δεν θα πρέπει να υπάρξει απομάκρυνση από τους βασικούς μας στόχους και πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο ε, μήνυμα ότι ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να διατυπωθεί το ταχύτερο δυνατόν, να είναι ουσιαστικός, οι κυρώσεις να είναι ουσιαστικές ε, επίσης ε, και δεν θα πρέπει απλά ε, να κάνουμε μια μεγάλη φασαρία στην αρχή και μετά τίποτα. Δεν χρειάζεται κανείς να χρησιμοποιεί την οδολογία του μαρξισμού για να προωθήσει τις απόψεις αυτές. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τους ενδιαμέσους, τους φορολογικούς συμβούλους, τους δικηγόρους, τις τράπεζες που πολλούν μηχανισμούς βελτιστοποίησης των φορολογικών υποχρεώσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ανταλλάξουμε σε επίπεδο πληροφορίας με τις φορολογικές αρχές της κάθε χώρας. Έτσι οι φορολογικές αρχές θα μπορέσουν να ανοιχνεύουν τις διοικητικές τους αδυναμίες και παραθυράκια. Και οι προτάσεις αυτές με τη σειρά τους θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά, διότι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς αυτούς, είτε επιχειρήσεις είτε ιδιώτες, θα είναι γνωστή από τις φορολογικές υπηρεσίες. Ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ έχει πολλά να πει και οι προτεραιότητές μας συμπίπτουν. Η, η, Επιτροπή θα επιμείνει σε αυτό. Ένα τρίτο, σημείο το οποίο θα ήθελα να ζητήσω την προσοχή σας. Ένα σημαντικό προϊόν των απατών στο ΦΠΑ τροφοδοτεί εγκληματικά δίκτυα και ένα τμήμα πηγαίνει και σε τρομοκρατικά δίκτυα. Ε, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες φύγονται από τις λεγόμενες απάτες τύπου γαϊτανάκι, καρουσέλ. Ε, πολλές φορές στείνονται από ε, εγκληματικές οργανώσεις. Σαν παράδειγμα, απάτες της ποσοστώσης του άνθρακα, 5 με δις ευρώ απώλειες για τα κρατη και η οργάνωση αυτή ε, κερδίζει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η απάτη για τα ΦΠΑ λοιπόν φύγει τον βασικό πόρο ε, των κρατών μελών, το VAT gap. Μπορούμε να πούμε ότι συνολικά υπολογίζεται σε 110 δις κατέτος, από τα οποία 40 με 60 είναι διασυνοριακές απάτες τα κενά στο σύστημα του ΦΠΑ έτσι όπως είναι σήμερα, ε, συνδυαζόμενο με πολλές διευκολύνσεις για την χρήση τραπεζικών λογαριασμών εκτός, ε, από την, εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ε, μειώνουν, λειτουργούν θα έλεγα αρνητικά για τα έσοδα από ΦΠΑ και επιτρέπουν στους απαταιώνες να εκμεταλλεύονται τα χρήματα αυτά αυτό το φαινόμενο το οποίο είναι τεκμηριωμένο τώρα πια πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε εμείς ε, την απάτη στο ΦΠΑ το διασυνοριακό σαν κάτι το μοιραίο. Έχουμε ένα μεταβατικό καθεστώς εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το 2013. Και έχει γίνει το προσωρινό μόνιμο θα έλεγα είναι κάτι το οποίο έχει προκληθεί από την ύπαρξη 28 διαφορετικών συστημάτων που επιτρέπουν τη λογική του καρουσέλ. Περιμένω λοιπόν την υποστήριξη του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις προτάσεις τις οποίες θα κάνουμε το ε, Φεβρουάριο, μάλλον το Φινόπορο, συγγνώμη, για να ενισχύσουμε τον αγώνα μας εναντίον αυτής της μεγάλης απάτης. Θα είναι ένα ισχυρό μέσο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, όπως έχουν δείξει ορισμένα ντοκιμοντέρ, ένα Ολλανδικό ντοκιμοντέρ ε, των τελευταίο μήνες έδειξε τη σχέση ανάμεσα σε, αυτές τις, σε αυτούς τους παράγοντες. Τέλος και θα τελειώσω εδώ Για την πρόσβαση στα έγγραφα είμαστε υπέρ της διαφάνειας και θα συνεργαστούμε μαζί σας. Εμείς εξετάζουμε τα αιτήματά σας για πρόσβαση σε έγγραφα με πολύ σοβαρότητα και έχουμε αφιερώσει πολλές δυνάμεις για να το πετύχουμε και να ανταποκριθούμε. 650 έγγραφα in camera και κλεισμένων των θυρών. 800 έγγραφα μέσω κλειστού δικτύου και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στο μέλλον. Ένα μεγάλο κομμάτι των εγγράφων του κώδικα συμπεριφορά μας ε, διαφεύγει και όπως είπε ο πρόεδρος η κατάσταση εδώ ίσως να είναι λίγο απογοητευτική. Ξέρω ότι δεν είσαστε ικανοποιημένοι. Να σας πω ότι στόχος μας είναι πράγματι να παράσχουμε στην Επιτροπή σας τα έγγραφα τα σχετικά με την εντολή που έχετε για τη δουλειά σας. Το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Η ομάδα ας πούμε συμπεριφοράς για τη φορολογία των επιχειρήσεων ασχολείται με πάρα πολλά θέματα. Λίγα από τα θέματα αυτά έχουν σχέση με τις δικές σας αρμοδιότητες. Ε, κάποια άλλα δεν χρειάζονται. Εγώ μάλιστα έστειλα μια επιστολή εξ ονόματος της Επιτροπής στο Συμβούλιο, έτσι ώστε κάθε θεσμικό όργανο και το Συμβούλιο δηλαδή να παρέχει πρόσβαση στα έγγραφά του. Έχουμε βέβαια όρια σε σχέση με το Συμβούλιο και θα τελειώσω εδώ, αλλά δεν θα πρέπει αυτό το πράγμα να το ξεχνάμε στα πλαίσια ε, της ε, πραγματικής προσπάθειας ε, και στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης ε, που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Ε, συναντήθηκε ο Γενικός Διευθυντής ε, με τους εισηγητές της Επιτροπής σας, τους συντονιστές της Επιτροπής σας και συνεχίζουμε την προσπάθεια. Αυτά είχα να σας πω εισαγωγικά, ζητώ συγγνώμη διότι μακρηγόρησα, αλλά έχουμε πάρα πολλά πράγματα μπροστά μας και δυστυχώς όπως είπα μίλησα περισσότερο από όσο έπρεπε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε. Ο Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ελπίζουμε και είμαστε πεπισμένοι ότι από κοινού, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστούμε αγαστά σε αυτά τα δύσκολα φορολογικά ζητήματα. Το βασικό μας πρόβλημα ποιο είναι. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε η προθυμία συνεργασίας της με το Κοινοβούλιο, αλλά κατά κύριο λόγο η απροθυμία, η διστακτικότητα, και το λέω μετριοπαθώς, κάποιων κρατών μελών που μπλοκάρουν. Και δεν αφορά μόνο το έγγραφο που σας έδειξα προηγουμένως, αλλά και ένα άλλο που αφορά τις ειδικές φορολογικές συμφωνίες, τα tax rulings. 11 είναι οι χώρες που έχουν τέτοιες ειδικές συμφωνίες και οι 11 χώρες, με μία εξαίρεξη, το Λουξεμβούργο, που δεν ε, αμαύρωσε τις ε, σελίδες, οι υπόλοιπε 10 μας έδειξαν μαύρα έγγραφα. Και σε μια περίπτωση που πρόκειται για ένα ομοσπονδιακό κράτο, αυτό αφορά μία περιφέρεια και μόνο και είναι μαύρο όλο το έγγραφο. Πού είναι η βούληση να δείξουμε διαφάνεια και να αυξηθεί η δημόσια πίεση για τις μεταρρυθμίσεις. Είναι μάλλον χαλαρή στα κράτη-μέλη. Και αυτό δεν είναι μόνο δυσπιστία προς το Κοινοβούλιο, η στάση αυτή που είναι το μόνο εκλεγμένο όργανο, αλλά αυτό δεν δικαιολογείται και από τη φορολογική αρμοδιότητα που έχουν τα κράτη-μέλη. Υποστηρίζουμε αυτά που είπατε ε, τα τρία ε, για το ΦΠΑ, για τους φορολογικούς παραδείσους και την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιριών επειδή έχουμε καθυστερήσει και αργότερα ξεκινήσαμε και λίγο περισσότερο μιλήσατε κι εσείς και καλά κάνατε, θα πρότεινα να αρχίσει αμέσως η συζήτηση με τους δύο συνεισηγητές ε, με τις ερωτήσεις και ξέρετε ότι μέχρι τις 10.30 έχουμε συνεδρίαση. Ο κύριος Σκόφουτ πρώτος και μετά ο επόμενος. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας βλέπουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα, αναφερθήκατε στην μάχη για την διαφάνεια και αυτή η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να σας βοηθήσει. Από κοινού μαζί με τα κράτη-μέλη, είτε πρόκειται με την ενοποιημένη φορολογική βάση για τις εταιρείες, είτε πρόκειται για την αναφορά αναχώρα, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η απαιτούμενη διαφάνεια θα γίνει ο κανόνας. Το ερώτημά μου λοιπόν συνδέεται με αυτό το ζήτημα, γιατί η Επιτροπή του Παναμά πρόσφατα βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί μάθαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να κάνουν αμοιβέ ανταλλαγέ σε πληροφορίες όταν πρόκειται για τι αναφορέ, για του κανόνε αναφορών. Έχουν στα χέρια του τα δεδομένα, αλλά δεν είναι διατεθειμένες να τα ανταλλάξουν. Είναι αυτή και η δική σα εκτίμηση και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Γιατί ένα από τα κριτήρια, όπως αναφέρατε πριν, για τους μαύρους καταλόγους των ε, φορολογικών παραδείσων είναι αυτές οι κοινέ αναφορές. Μπορούμε λοιπόν να, να μάθουμε ποια είναι η αντίδραση της Επιτροπής για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Σε ό,τι αφορά τη λίστα τώρα που, στην οποία αναφερθήκατε ως βασική προτεραιότητα, την μαύρη αυτή λίστα, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο ότι λείπουν μερικά κριτήρια από την λίστα αυτή. Μπορείτε όμως να μας δώσετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Και τέλος, αναφερθήκατε στον ε, κώδικα διοντολογίας ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή από το 1998. Υπάρχει ίσως η σκέψη να επανεξετάσει λίγο η Επιτροπή την ομάδα αυτή, την, την εντολή λειτουργίας ομάδας αυτής, σε ό,τι αφορά τη, τα διασυνοριακά φορολογικά καθεστώτα, πόσο αποτελεσματικά είναι. Αναφερθήκατε στην ενιαία αγορά, αναφερθήκατε στην ενοποιημένη φορολογική βάση για τις εταιρείε. Εδώ όμως θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε από κοντά τον κώδικα διοντολογίας και να δούμε αν υπάρχουν κάποιες νέες προοπτικές, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε στο μέλλον σε σχέση με τον κώδικα αυτό. Ευχαριστώ κύριος Επίτροπος. Παρακαλώ να τηρούμε το πεντάλεπτο. Okay. Um, first, I'm, I'm pleased. Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρόοδο σε ό,τι αφορά το Juris. Πιστεύω ότι είναι απόλυτα εναρμονισμένο με αυτό που είχαμε οραματιστεί στην αρχή σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες δικαιοδοσίες τις οποίες ελέγξαμε αλλά και τις διαδικασίες ελέγχου που διεξάγουμε. Υπάρχουν ομάδες ειδημόνων από κράτη-μέλη και από την Επιτροπή έχουν ε, ξεκινήσει ήδη από τον ε, Μάρτιο να εξετάζουν τις περιοχές αυτές. Δευτερευόντως, ομάδες οι δημόνων θα εξετάσουν τις πληροφορίες αυτές, θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές και μέχρι τον ε, Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η δουλειά τους και επόμενο βήμα αναμένεται να είναι ότι η λίστα αυτή θα παρουσιαστεί στην ΕΚΟΦΗΝ μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Θα μπορέσουμε ίσως να έχουμε και μέτρα σε ό,τι αφορά τις χώρες αυτές που θα βρίσκονται στη λίστα. Παραμένουμε αισιόδοξοι και έχουμε, μας χαροποιεί ιδιαίτερα ο ενθουσιασμός των κρατών μελών να συμμετάσχουν στην διαδικασία αυτή σε ό,τι αφορά τώρα τις Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν αμοιβαιότητα σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι απόλυτα εναρμονισμένες με την παγκόσμια ανταλλαγή πληροφοριών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν την ευθύνη να, να ακολουθήσουν τους κανόνες ό,τι αφορά την παγκόσμια προσπάθεια εναντίον της ε, φοροδιαφυγής και πρέπει να προσαρμόσουν το σύστημά τους. Υπάρχει ένα ευρύ φέσμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και, και την Ευρωπαϊκή Ένωση να δουλέψουν από κοινού, να έχουν επικοδομητικές συνομιλίες. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει με όλα αυτά τα δεδομένα η, η νέα διοίκηση, η νέα κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, διοντολογία και την ε, φορολογία των εταιριών, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να εξασφαλίσουμε δίκαιη φορολόγηση, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε κακές φορολογικές πρακτικές. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανάγκη μεταρρύθμισης του κώδικα αυτού διοντολογίας, ναι, βεβαίως είναι κάτι που γίνεται όλο και πιο εμφανές. Αυτή η Επιτροπή και αυτό το Κοινοβούλιο έχει επαναλάβει αρκετές φορές ότι είμαστε έτοιμοι να, να εργαστούμε από κοινού με τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να μεταρρυθμίσουμε τον κώδικα αυτό, να τον κάνουμε πιο αποτελεσματικό και πιο δίκαιο. Και θα ήμασταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι να βοηθήσουμε στην ε, διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Γιάτσεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λοιπόν, αυτό που θα με ενδιαφέρει κύριε Επίτροπε είναι να μάθω πώς αξιολογείτε την υλοποίηση από πλευράς κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στους τομείς που συζητούμε. Έχετε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντά σας για να ενισχυθεί αυτή η εφαρμογή της νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη. Έχει τους απαραίτητους πόρους στη διάθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίζει τη σωστή επιβολή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Αυτή ήταν η πρώτη μου ενότητα ερωτήσεων. Και στη συνέχεια θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο την πρωτοβουλία για τη ρύθμιση των φορολογικών συμβούλων, φοροτεχνικών. Προετοιμάζεται και άλλα τέτοια κείμενα στο προσεχές μέλλον. Ή και στο απότερο. Και τέλος, το 2013 ξέρετε μια επιστολή με τους άλλους ομολόγους σας τότε ε, υπουργού Οικονομικών των κρατών μελών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να υπάρξει ένα αντίστοιχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αμερικανική ΦΑΤΚΑ. Εκεί υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές που έχετε εντοπίσει, γιατί αυτό το αμερικανικό εργαλείο στι ΗΠΑ είναι αρκετά βαρύ, αλλά και αρκετά αποτελεσματικό ταυτόχρονα. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο και ευχαριστώ τον συνάδελφο για τι ερωτήσει. Ευχαριστώ. Έδωσα εντολή στι υπηρεσίες μου, όπως μου ζητήσατε, να μελετήσουν ε, εάν έχει γίνει έγκαιρη και σωστή μεταφορά ε, της νέας ε, νομοθεσίας των οδηγιών για τη διαφάνεια και κατά της φοροδιαφυγής. Και σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη δεν απάντησαν, κινήσαμε τη διαδικασία επί παραβάση. Το πρώτο στάδιο είναι ε, οι επιστολές, οι προδιοποιητικές. Σε 39 περιπτώσεις, δεν θα τις αναφέρω όλες αναλυτικά, έχετε ε, την πληροφόρηση. Τα περισσότερα κράτη-μέλη μετά την προειδοποίηση που του στείλαμε κοινοποίησαν ε, τη μεταφορά της νομοθεσίας. Ε, ωστόσο υπάρχουν 12 κράτη-μέλη για τα οποία κρεμούν ακόμα κάποιες δράσεις. Μετά από αυτό το πρώτο έλεγχο πληρότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα εξετάζει κατά πόσο εφαρμόζονται και μεταφέρονται σωστά οι οδηγίες στο εθνικό δίκαιο για το ΤΑΚΟΑΝ σε έξι κράτη-μέλη. Είχαμε ερωτήματα σε σχέση με τη συμμόρφωση για περιπτώσεις που τώρα έχουν κλείσει. Και πάλι τις λεπτομέρειες τις έχετε στη διάθεσή σας αν θέλετε. Για την ΤΑΚ 2 ε, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αξιολόγηση και ελπίζουμε να είναι λίγες οι παραβάσεις. Όπως βλέπετε, εμείς επιδεικνύουμε τη δέουσα επιμέλεια και αποδίδει αυτό, γιατί τα κράτη-μέλη τείνουν να προσαρμόζουν με ταχύς ρυθμούς τη νομοθεσία τους στα δικά μας αιτήματα. Έχετε τις ε, πληροφορίες αυτές και μιλώ υπό τον έλεγχό σας. Το τελευταίο που με ρωτήσετε, τη τελευταία διετία, έχουν γίνει πολλά σε σχέση με τους ε, Φορολογικού συμβούλου, φοροτεχνικού, για να καταπολεμούμε αποτελεσματικά τη φοροαποφυγή και τη διαφυγή. Τώρα όμως θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και την κατάσταση εκείνων που ε, διαφημίζουν και προβάλλουν την ε, φοροαποφυγή με τη φορολογική βελτιστοποίηση, με ανθρώπους πάρα πολύ ειδικού που γνωρίζουν όλους τους ε, νόμους, τους δρόμους, τις δυνατότητες που έχουν πάρα πολύ καλά και να δούμε τι εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκεί. Αυτό που χρειάζεται τώρα λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτές ακριβώς τις πρακτικές. Τρία κράτη-μέλη έχουν υποχρεώσει με την νομοθεσία τους να ε, δημοσιεύονται ε, αυτά τα σχήματα φορολογικής βελτιστοποίησης πριν την εφαρμογή τους. Και μπορώ να υπολογίζω και στη βοήθεια τη δική σας ε, για να υλοποιηθούν όλα αυτά το συντομότερο και μάλιστα πριν το θέρος. Για τη ΦΑΤΚΑ τώρα εφαρμόζεται σε διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατηθειμένη να συνεχίσει τον παγκόσμιο διάλογο που γίνεται με τρίτες χώρες για να είμαστε και πιο αυστηροί απέναντι σε μη συνεργαζόμενες χώρες. Καλώς, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Βέβαια, μας μας ενδιαφέρει να ακούσουμε και ποιες είναι οι χώρες αυτές. Ακριβώς. Που έχουν προχωρήσει σε λήψη μέτρων και νομοθεσία για τους μεσάζοντες και τους φορολογικούς συμβούλους. Ο καθηγητή Ντάριου Ρωσάτη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, γιατί ακολουθούν τώρα μιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τι πληροφορίε τι οποίε μα δίνετε. Δύο ερωτήσει. Η πρώτη για τα εξαρτώμενα λεγόμενα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε μια ακρόαση στις αρχές της εβδομάδας γύρω από αυτό και από ό,τι φαίνεται κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι δεν ελέγχουν πλήρως τις ρυθμίσεις των λεγόμενων εξαρτημένων εδαφών και στα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης αλλά και εκτός αυτής. Αυτό αφορά ε, τις ε, νήσους της Μάνχης, τις νήσους της Καραϊβικής, που ανήκουν ή ελέγχονται από την Ολλανδία, από τα Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Γαλλία κτλ. Θα ήθελα να μάθω αν πράγματι συνειδητοποιείται το ότι υπάρχει μια διαδικασία μεταφοράς των κερδών προς τα εδάφη αυτά για φορολογικούς λόγους σε μεγάλη κλίμακα στην Ευρώπη. Και τι μπορούμε εμείς να κάνουμε έτσι ώστε να αναγκάσουμε τα κράτη-μέλη που εμπλέκονται να προσπαθήσουν να, πάρουν τις, να κάνουν τις απαιτούμενες νομικές αλλαγές έτσι ώστε να μην υπάρχουν αναντιστοιχίες στις νομοθετικές ρυθμίσεις μεταξύ των εδαφών που ανήκουν μένα επίσημα στο ίδιο κράτος μέλος και εν μέρει ανήκουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να κάνουμε κάτι λοιπόν με αυτό ή θα πρέπει να ανεχθούμε αυτή την κατάσταση. Και η δεύτερη ερώτησή μου, σύντομα, η τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου σχετικά με τα δημόσια CBCR Κάποιοι αντέδρασαν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασαν τις ανησυχίες τους ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να οδηγήσει στη δημοσιοποίηση εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων και μπορεί αυτό να έχει δύο συνέπειες για τις χώρες αυτές. Η πρώτη συνέπεια είναι ότι οι θυγατρικές μη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα αντικατασταθούν, θα απομακρυνθούν, θα μετακινηθούν σε άλλες χώρες. Και η ροή των επενδύσεων θα στερεύσει και θα πάει προς τις Ηνωμένε Πολιτείες και τον Καναδά. Η δεύτερη πιθανή συνέπεια είναι ότι μπορεί να υπονομεύει τα επίπεδα του ΟΣΑ. BEPS 13 σαν παράδειγμα, BEPS δράση 13, και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί οι χώρες μέλη να το χρησιμοποιήσουν ως άλοθη για να μην γίνει σεβαστή η συμφωνία. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενήμερη αυτών των ανησυχιών. Ευχαριστώ κύριε ε, Ρωσάτη. Το τελευταίο αυτό είναι στην νομοθετική διαδικασία. Την περασμένη εβδομάδα κάναμε και ακρόαση. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Euh. Πολλές ερωτήσεις, λίγος χρόνος για να απαντήσω. Θα προσπαθήσω όμως να το κάνω τηλεγραφικά για την πρώτη σας ερώτηση. Συνειδητοποιούμε τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Αυτό ανήκει και στην διαδικασία του listing και στα πλαίσια επίσης του κώδικα συμπεριφορών εμείς θα πρέπει να εξετάσουμε με συγκεκριμένο τρόπο ε, κάποιες δικαιοδοσίες όπως το Jersey, το Guernsey, την ίσο του Μαν ε, που έχουν εξαιρεθεί από τις εργασίες ε, του κώδικα αλλά θα πρέπει τα παγκόσμια στάνταρς για την διαφάνεια να γίνονται σεβαστά. Σχετικά τώρα με το CBCR δημόσιο κομμάτι υπάρχουν δύο θέματα. Υπάρχει το θέμα της, ε, ρύθμισης αν θέλετε. Εμείς εδώ προτείνουμε δημοσιοποίηση, διαφάνεια. Ε, προσθέτοντας επίσης και την δυνατότητα έκφρασης αντίθεσης μάλλον ανάμεσα στη διαφάνεια και την επένδυση όπως επίσης και την αρχή της αμοιβαιότητας με τις ΗΠΑ. Ε, αυτό είναι κάτι που συζητώ με τον Άγχελ Γκουρία του ΩΣΑ. Ε, θα πρέπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε αυτό. Είμαι όμως πεπισμένος ότι στα πλαίσια κάποιων ορίων τα οποία σεβαστήκαμε στην πρότασή μας, δεν υπάρχουν εσωτερικές αντιφάσεις και νομίζουμε ότι η διαφάνεια θα επικρατήσει. Αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το αποφασίσουν αυτό. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσει τον σεβασμό των ιδίων του των θέσεων ε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνένεση στην ιδέα της διαφάνειας, δεν θα εγκαταλείψουμε τη μάχη, αν και οι συζητήσεις που βρίσκονται σε προκατακτική φάση στο Συμβούλιο δείχνουν ότι ο αγώνας θα είναι σκληρός. Πάντως εμείς σαν Επιτροπή είμαστε υπέρ της δημοσιοποίησης των εκθέσεων αναχώρα. Μάλιστα εγκρίναμε, μάλλον ελέγξαμε και τις τροπολογίες και καταλάβαμε και στο Κοινοβούλιο θα υπάρξει δυσκολία εξέβρεση κοινή γραμμή για αυτό το θέμα. Και ο προσανατολισμός της διατάξης BEPS είναι σημαντικός για τη διάβρωση της ε, βάσης και μεταφορά των κερδών. Για τις χώρες που δεν συνεργάζονται, είναι 33 οι δικαιοδοσίε των κρατών μελών, εδάφη των κρατών μελών, δεν είναι μόνο τα νησιά της Μάχης είναι ύποπτα <laughs> ω φορολογική παράδειση. Τα είπε και ο συνάδελφο αυτά και παρακαλώ να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά. Ο συνάδελφος Πολ Τάγκ των Σοσιαλδημοκρατών. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Μοσκοβισή, που είστε εδώ. Εχθέ ήταν η πρώτη ακρόαση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε τη συζήτηση για την ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιριών. Και ένα μέρος της συζήτησης, όπως άκουσα και από εσά, ήταν ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η απάντηση της Ευρώπης, μια πιο συντονισμένη δράση, σε ό,τι αφορά τις ε, προτάσεις ε, φορολογίας της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία μείωσε τη φορολογία σε 15%. ξεκινώντας ένα σύστημα που δεν είναι παραδοσιακά αμερικάνικο, έχει να κάνει περισσότερο με τις διαφορετικές περιοχές. Πώς λοιπόν κρίνεται αυτήν την δράση της Αμερικανικής κυβέρνησης και τι πιστεύετε σε ό,τι αφορά την ενοποιημένη, φορολογική, την ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιριών. Η δεύτερη ερώτησή μου, τι βλέπετε να συμβαίνει στα διαφορετικά κράτη-μέλη, γιατί ο όσα ανέφερε νομίζω 12 α, χώρες οι οποίες θα πρέπει να αποκαλύψουν πληροφορίες. Βλέπετε κάποια πρωτοβουλία από πλευρά των κρατών αυτών. Γιατί πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτή μπορεί να είναι η στιγμή που θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Αυτό το θέμα των φορολογικών συμβούλων είναι πραγματικά φλέγον γιατί από τα 403 έγγραφα ε, τα 100 και πλέον ε, αφορούσαν τράπεζες και μόνο το ένα έγγραφο αφορούσε φορολογικούς συμβούλους ή φοροτεχνικούς. Επίτροπος. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας εφησυχάσω εδώ ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ένας από τους ε, βασικότερους εταίρους μας στη μάχη αυτή και αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε μόνο και μόνο γιατί έγιναν κάποιες προσαρμογές. Όπως σας είπα, ήμουν δύο εβδομάδες πριν στις Ηνωμένε Πολιτείε, μίλησα με αρκετούς ε, ηγέτες εκεί μεταξύ των οποίων την Κριστιαν ε, Λαγκάρ, τον Γκάρικον, και το μήνυμα που τους πέρασα ήταν ότι η Επιτροπή έχει πάντοτε κατά νου το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά τα φορολογικά ζητήματα. Την προηγούμενη εβδομάδα οι Ηνωμένε Πολιτείες ανακοίνωσαν κάποιες μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά την φορολογία των εταιριών η φορολογία τους παραμένει στο 39% αρκετά παραπάνω από την φορολογία εταιριών που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι εταίροι παραμένουμε συντονισμένοι στην προσπάθειά μας να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως θα ξεκινήσουμε, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και πιστεύω ότι δεν ε, ε, υλοποιήθηκε το, το χειρότερο σενάριο που είχαμε κατά νου. Αλλά είναι ανάγκη να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε από κοντά. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα δυναμικό περιβάλλον σε ό,τι αφορά την φορολογία των εταιριών. Και η καλύτερη δράση που μπορούμε να έχουμε είναι να εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα BEPS μέχρι το 2020 μαζί με τους εταίρους μας των ΩΣΑ και βεβαίως να προωθήσουμε το CCTB. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτή την ανάγκη σταθερότητας σε ό,τι αφορά τις φορολογικές βάσεις. Είμαστε ε, έτοιμοι να κάνουμε μια πρόταση τον Ιούνιο σε ό,τι αφορά τους διαμεσολαβητές. Τώρα δεν ξέρω αν θα πρόκειται για κυρώσεις για αυτούς που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσωπική μου οπτική γωνία, όπως ξέρετε, είναι υπέρ τέτοιων κυρώσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούκα από την ομάδα Ισία, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ένα ουσιαστικό στοιχείο στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και της δικής μας Επιτροπής στην καταπολέμηση του ξεπλήματος ε, χρήματος και της φοροδιαφυγής είναι η βελτίωση της ενημέρωσης που έχει το δημόσιο με μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερες απαιτήσει, μητρώα κλπ. Αλλά κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι να μπορούν τα κράτη να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες, να τις διεκπαιρεώνουν, να έχουν τους απαραίτητους πόρους. Τώρα με τις εργασίες της δικής μας Επιτροπής, αλλά και προσωπικά με κάποιες επαφές που είχα, έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει αυτό το δυναμικό. Ε, ξέρω από πολλά κράτη-μέλη ότι Υπάρχουν κάποιες ύποπτες περιπτώσεις και, και οι οποίες δηλώνονται ε, με τους ισχύοντες κανόνες μόλις το 1% ε, μπορούν να διαχειριστούν οι αρμόδιες αρχές που μπορεί να είναι η εφορία, μπορεί να είναι η εισαγγελία, διοκτικές αρχές κτλ. Δηλαδή αν υπάρχει υποψία και μόνο, ο ύποπτος έχει πιθανότητα 99% να μην πάθει τίποτα. Γιατί δεν υπάρχουν οι πόροι για να μπορούν να τα επεξεργαστούν αυτά τα κράτη. Άρα αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει μια αντίφαση. Από τη μια εμείς υποθέτουμε ότι με εγκληματικές δραστηριότητες ε, χάνει 3 εκατομμύρια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ε, τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να αφιερώσουν τους απαραίτητους πόρους ε, στην αποκάλυψη και δίωξη. Και μιλώ και για ανθρώπινο δυναμικό και για υλικοτεχνικό. Κανονικά αυτό θα πρέπει να αυτοχρηματοδοτείται και πολύ άνετα από τα έσοδα που χάνουν τα κράτη. Ε, το αναγνωρίζετε αυτό ως αντίφαση. Πώς το δικαιολογείτε και τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είναι κατάφοροι ε, πώς να το πω, αδράνεια σε περίπτωση τέτοιων ε, καταστάσεων. Ευχαριστώ κύριε Λούκο, ο Επίτροπος. Με χαρά διαπιστώνω ότι συμφωνούμε, που δεν συμβαίνει πάντα κύριε Λούκο. Ε, και είναι προφανής απόλυτη ανάγκη καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Αυτή η κοινή διαπίστωση είναι κάτι ε, στο οποίο καταλήγουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Και συμφωνούμε ότι η Ευρώπη σε αυτό το θέμα δεν είναι μόνο απαραίτητη αλλά και χρήσιμη. Αυτή η Ευρώπη που ορισμένοι την επικρίνουν καμιά φορά. Κατά τα άλλα αυτό είναι και τμήμα του ευρωπαϊκού αφηγήματο που θα πρέπει εμεί να προωθούμε και να προβάλλουμε και να υπερασπιζόμαστε περισσότερο απέναντι στους πολίτε γιατί εδώ είναι απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί να δράσει. Είναι υπαρκτό αυτό το πρόβλημα στο οποίο αναφέρεστε και χρειάζονται και πραγματικές απαντήσεις. Αλλά να μην υπερβάλλουμε σε προηγούμενη ιδιότητά μου, πριν αναλάβω επίτροπος, ήμουν δύο χρόνια υπουργό Οικονομικό τη Γαλλίας. Και μπορώ να σας πω ότι ο υπουργό οικονομικός για μια σειρά από λόγου θέλει να αρχίσει διάφορα προγράμματα καταπολέμησης και οικονομικούς λόγους και ηθικούς και πολιτικούς και άλλους, γιατί είναι έσοδα για το κράτος, για να μειώνονται τα ελλείμματα, που είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Και στην περίπτωση της Γαλλίας κάθε χρόνο εμείς, καλά εγώ δεν είμαι πλέον εκεί, εμείς οι Γάλλοι εννοώ, έχουμε προγράμματα για να συλλέγουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια φόρους ε, από τη φοροδιαφυγή και την φοροδιαφυγή. Έχετε δίκιο, παρόλο που τα ποσοστά που δώσετε θεωρώ πάρα πολύ υπερβολικά. Ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη ε, για να δημιουργούνται όταν χρειάζονται ή να βελτιώνονται όταν χρειάζονται οι διοικητικές ικανότητές τους και δυνατότητες για να είναι ακόμα πιο αποτελεσματική αυτή η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Κάνουμε και εργαστήρια τα οποία χρηματοδοτούνται από διάφορα προγράμματα για τη φορολογία και με μηχανογράφηση και με έλεγχο των νέων τεχνολογιών που είναι πάρα πολύ σημαντικές φυσικά για να αντιμετωπίζονται αυτές οι περιπτώσεις. Πάντως συμφωνώ ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουν τα κράτη-μέλη ότι δεν είναι μόνο καθήκον τους, αλλά και προς το συμφέρον τους να έχουν αυτή την διοικητική ικανότητα για να συλλέγουν περισσότερους φόρους και να καταπολεμούν καλύτερα τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Με χαρά υιοθετώ αυτό το μήνυμα, να το διαβιβάσω στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Υποθέτω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τα στοιχεία στα χέρια της ε, για τις ε, δυνατότητες των κρατών μελών. Πώς θα μπορούσατε να μας τα διαβιβάσετε και αυτά. Από τους φιλελευθέρους, η Μάιτε Ρουίθ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Μοσκοβισή, χαίρομαι πάρα πολύ που μας λέτε ότι τα 160 δισεκατομμύρια ευρώ φόρο διαφυγής ετησίως ε, δεν μπορούν να θεωρηθούν ε, κάτι το ε, δεδομένο και νομοτέλεια. Και θα πρέπει να έχει και πολιτικές επιπτώσεις και πολιτικές ευθύνες η αδράνεια. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπατε. Να επανέλθω λίγο στις κτίσεις και τα εδάφη που εξαρτώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 200.000 εταιρείε ε, ε, είχε η Μόνσα Φωσέκα στα έγγραφα του Πάναμα και οι μισές ήταν στις Βρετανικές νήσους. Είπατε ότι θα τα κοιτάξετε. Στις Βρετανικές Παρθένες νήσους. Αλλά αν δεν μπορεί το κοινοτικό κεκτημένο να εφαρμόζεται με άμεσο τρόπο σε αυτές τις κτήσεις των κρατών μελών, εσείς ποιε αρμοδιότητες έχετε ουσιαστικά. Εντάξει, να το κοιτάξετε, να το κοιτάξετε και πού θα πάμε, πού θα καταλήξουμε. Δεν είναι αποτελεσματικό αυτό. Χρειάζεται αλλαγή των συνθηκών. μιλήσατε για κάποια προθυμία για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών. Θα μπορούσατε να μας το εξηγήσετε, να μας δώσετε λίγες ε, περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί λέτε ορισμένες από αυτές τις, ε, τους δισταγμούς μάλλον που έχουν τα κράτη-μέλη δικαιολογούνται και άλλοι πάλι όχι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Επίτροπος, παρακαλώ. Τώρα έχετε και λίγο περισσότερο χρόνο, θέλετε. Η απάντηση είναι απλή, παρότι έχω χρόνο περισσότερο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία έχει δύο αν θέλετε κλάδους. Ή μιλάμε για εδάφη τα οποία είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί ε, σε σχέση με τη διαδικασία του listing, εμείς πραγματικά αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι να γίνει σεβαστό το χρονοδιάγραμμα και το επαναλαμβάνω αυτό με αφορμή την ερώτησή σας. Είμαι ικανοποιημένος αρκετά για τον τρόπο που έχουμε προχωρήσει μέχρι τώρα και σχετικά αισιόδοξο γιατί μπορούμε να έχουμε αυτή την πανευρωπαϊκή λίστα των φορολογικών παραδείσων με τις επακολουθούμενες ακυρώσεις. Τώρα, στην άλλη περίπτωση, αν είναι εδάφη μέσα στην Ένωση, που έχουν ένα διαφορετικό καθεστώς ανάλογα με τις ρυθμίσεις της κάθε χώρας. Σε αυτή την περίπτωση το κοινό και εκτιμένο, το κοινοτικό, είναι αυτό το οποίο επιβάλλει τους κανόνες του. Η κατάσταση ίσως θα επιβαρυνθεί όταν μια μεγάλη χώρα αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να εξετάσουμε στη διαδικασία να διαβεβαιώσω ότι οι ενδιάμεσοι που δραστηριοποιούνται στα εδάφια αυτά θα καλυφθούν από την επόμενη πρότασή μας γιατί δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν παραθυράκια τα οποία να επιτρέψουν να υπάρξει στρεβλή χρήση της δυνατότητας αυτής. Ο Μικέλ Ουρμπάν από την Eh, Ευχαριστώ Επίτροπε. Επτά εκπρόσωποι της BNP και ε, τρεις εκπρόσωποι άλλης τράπεζας έχουν καπιτάλες. Σάταντερ έχουν κρατηθεί στα πλαίσια των αποκαλύψεων της λίστας Φαλσιανή το θέμα το τι κάνουν όλοι αυτοί οι σύμβουλοι, τα διοικητικά σελέχη και τα λοιπά, ο ρόλος τους είναι πάρα πολύ μεγάλος για τις φορολογικές διευκολύνσεις οι οποίες ισχύουν ε, για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η συνενοχή των ενδιαμέσων αυτών είναι προφανής και διαρωτώ με αν θα πάρετε μέτρα στον τομέα αυτό ε, τα μέτρα αυτά θα είναι διακοσμητικά ή θα πηγαίνουν στη ρίζα του, του προβλήματος. Οι πολίτες ανησυχούν. Περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά βλέπουν ότι δεν έγιναν και πολλά πράγματα σε περιπτώσεις όπως τα LuxLeak, τα, οι περιπτώσεις του κυρίου Κανιέτε γύρω από τα Panama Papers και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις Λοιπόν, οι ενδιάμεσοι αυτοί, οι διαμεσολαβητές, τι είναι ρόλο παίζουν στην διαδικασία αυτή και τι κυρώσεις προβλέπονται, σαν παράδειγμα αφαίρεση επαγγελματικής άδειας δραστηριότητας, γνωρίζοντας και τον διεθνικό χαρακτήρα, η διαδικασία επίβλεψης ε, σε ποιον θα ανήκει. Θα ανήκει στις ευρωπαϊκές αρχές η εποπτεία ή στα κράτη-μέλη και τις αρμόδιες αρχές εποπτείας. Νομίζω ότι μήπως θα πρέπει να ζητήσουμε να υπάρξει ένας κατάλογος των δράσεων οι οποίες θα πρέπει να θεωρηθούν ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον συγκεκριμένο τρόπο. Παρακαλώ. Ορίστε, είπατε ότι θα τα διαβιβάσετε αυτά, τώρα σας ε, καλούν και συγκεκριμένα. Εξορισμού όταν μια οδηγία δεν έχει ακόμα κατατεθεί ε, στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Εγώ δεν μπορώ να τα αποκαλύψω αυτά εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απλώς και παρόλα αυτά η δράση μας ακριβώς επί των ενδιαμέσων για τα φορολογικά ζητήματα είναι ε, ότι συμφωνούμε ε, μαζί σας. Και έχει πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ζήτημα αυτό. Είναι ε, κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και επειδή γνωρίζουν τα θέματα αυτά τα νομικά, τα χρηματοοικονομικά, ε, ενθαρρύνουν την φοροαποφυγή και μάλιστα την υποβοηθούν. Χρειάζεται ένα πραγματικό σύστημα διαφάνειας και κινήτρων. Νομίζω θα ξανάρθω στην Επιτροπή σας ε, θα σας δώσω όλες τις προφορίες που θέλετε σε λεπτομέρειες και τα άλλα που μου ζητήσατε για τις ε, χώρες. Θέλω να σας αναφέρω τρεις αρχές επί των οποίων εργαζόμαστε με τη Γενική Διεύθυνση Τάξιουτ. Πρώτον, εμείς θα αντιμετωπίσουμε όλους τους ενδιαμέσους. Δεν θα περιοριστούμε σε ορισμένα επαγγέλματα. Όλα τα επαγγέλματα θα πρέπει να εξεταστούν και να τους αφορά. Δεύτερον, η πρότασή μας θα αφορά επίσης όλα τα σχήματα και τους μηχανισμούς φορολογικής βελτιστοποίησης. Δεν θα έχουμε εξαντλητικό κατάλογο μεν, ε, αλλά και αυτό είναι καλύτερο, γιατί επιτρέπει να προσαρμοζόμαστε. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, μηχανισμοί που κατασκευάζονται λόγω της τεχνογνωσίας και της οικονομικής και της ε, νομικής και εξελίσσονται αυτά. Και η τρίτη πρόταση θα έχει ε, στόχο όλα ε, τα κράτη. Αν οι ενδιάμεσοι εδρεύουν σε μια τρίτη χώρα και δεν πληρούν αυτές τις υποθέσεις, θα πρέπει ο φορολογούμενος να επομιστεί με την προσπάθεια αυτή αυτοί είναι οι τρεις άξονες επί των οποίων εργαζόμαστε και βεβαίως το θέμα των κυρώσεων τίθεται επίσης. Ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση αυτή. Είναι ευρύτατη πρόταση. Αν μπορώ να το πω αυτό από τώρα. Η κυρία Εύα Ζολή των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Περιμένω με μεγάλη ανημομονησία την πρόταση της Επιτροπή σε ό,τι αφορά τους ενδιάμεσους. Γνωρίζουμε το ρόλο που παίζουν. Η Επιτροπή Πανά εξετάζει όλους αυτούς τους ενδιάμεσους την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα και αναρωτιέμαι αν στην πρότασή σας θα προβλέπετε θα προβλέπονται ποινικέ κυρώσεις. σε ό,τι αφορά την, ε, την συμμετοχή τους για την ε, φοροδιαφυγή των ε, πελατών τους. Γιατί πιστεύω ότι ο ποινικό κώδικας σε κάποιες χώρες δεν είναι έτσι όπως θα πρέπει να είναι και ίσως είναι ανάγκη να το συζητήσουμε. Και μια δεύτερη ερώτηση. Μαθαίνουμε μεγάλη χαρά ότι σήμερα το απόγευμα η Επιτροπή, με συγχωρείτε η Επιτροπή σας απέτρεψε την απώλεια ενός ε, εκατομμυρίου, ενός δισεκατομμυρίου συγχωρείτε. Ποια ήταν λοιπόν η διαδικασία που ακολουθήσατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε. Ε, κύριος Επίτροπος. Δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά τους ενδιάμεσους, λοιπόν, είναι σημαντικό ο ορισμός των ενδιάμεσος να καλύπτει όλους αυτούς που προσφέρουν αυτές τις επιρεσίες, κατηγορίες επαγγελμάτων. Γιατί διαφορετικά υπάρχουν κενά στην, στις διαδικασίες που ακολουθούμε, αν δεν καλύπτουμε ένα ευρύ χάσμα ενδιάμεσων. σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει όταν πρόκειται για μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η Επιτροπή ε, προτιμά τον hard law αντί για τον soft law. Επομένως, λοιπόν, ακολουθούμε αυτήν την γραμμή. Σε ό,τι αφορά τους ενδιάμεσους, λοιπόν, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν ε, διαφάνεια σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, δεν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν ποινικέ κυρώσει. Σε ό,τι αφορά τι αποκαλύψεις που αναφέρατε της Εφημερίδα σουά δεν διάβασα την εφημερίδα, επομένω δεν έχω λεπτομέρειες. Θα τη διαβάσω στη συνέχεια. Απλά σας λέω ότι ότι πρόκειται η Τράπεζα Επενδύσεων και BERT είναι υπεύθυνοι αυτή οργανισμοί. Πρέπει να είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση σε ό,τι αφορά την χρήση των Ευρωπαϊκών Ταμείων είναι προσωπική μου φιλοδοξία ως επίτροπος να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Θεωρώ ότι όταν κανείς θέλει να είναι ηγέτης πρέπει να ηγείται με το παράδειγμα. Πάντοτε λοιπόν θεωρούμε ότι οι περιοχές που παίρνουν πόρους από, το, από τα ευρωπαϊκά ταμεία θα πρέπει να σέβονται τους φορολογικούς κανόνες. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από την δική σας βοήθεια για να έχουμε καλύτερη διαχείριση, ιδίως ό,τι αφορά τους ε, χρηματοοικονομικούς κανόνες. Σας ευχαριστώ λοιπόν που θίξατε το ζήτημα αυτό που μου επέτρεψε να σας παρουσιάσω αυτήν τη θέση σε ό,τι αφορά την ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω εκπρόσωπο της ομάδας EFTT. Οπότε το λόγο έχει η κυρία Μπάρμπαρα Κάπελ από την ομάδα ENF. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε Μοσκοβισή, που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας. Ε, θέλω να σας αναφέρω δύο τομείς ε, και να σας κάνω ερώτηση. Το ένα αφορά τις φορολογικούς παραδείσους και τη μαύρη λίστα και το δεύτερο τη φορολογική δικαιοσύνη. Είπατε σήμερα ότι η μαύρη λίστα θα πρέπει να έρθει μέχρι τα τέλη του έτους και είναι και δική σας προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είστε πεπισμένος ότι και το ΕΚΟΦΗΝ μέχρι το τέλος του έτους θα συμφωνήσει να καταρτιστεί ένας τέτοιος κατάλογος. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Πλην όμως έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν ακόμα κάποια προβλήματα ως προς τον ορισμό των κριτηρίων με τα οποία θα καταρτιστεί ο κατάλογος αυτό. Υπάρχουν κριτήρια του ΩΣΑ και κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι ο φορολογικός συντελεστής, η διαφάνεια, διεθνή συνεργασία ή προθυμία με την κοινωνία των κρατών. Και υπάρχει και ο κατάλογος 25 σημείων του FATF. Επίσης, στη συζήτηση για την οδηγία κατά του ξεπλήματος ε, χρήματος την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή ΕΚΟΝ αναφέρθηκε για ποιο λόγο δεν συμπεριλαμβάνεται ο Παναμάς ε, σε αυτή τη λίστα. Ποια είναι τα κριτήρια για τους υποψηφίους ή τις ενδεχομένως υποψήφιες χώρες που μπορεί να μπουν μπορεί και να μην μπουν στον κατάλογο αυτό. Και η έκθεση αναχώρα το συζητάτε αυτό ε, για, για τη συγκεκριμένη λίστα ή για όλες τις χώρες. Και μπορεί να υπάρχει αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Δηλαδή θα κληθεί ο Παναμάς να αποδείξει ότι τηρεί τους κανόνες. Υπάρχει μια έκθεση της Μαλτέζικης Προεδρίας για τη φορολογική δικαιοσύνη που λέει πάνω κάτω τα εξή και έχει υποβληθεί και στο ΕΚΟΦΗΝ της 7ης-8ης Απριλίου ότι χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων αλλαγών που γίνονται στη νομοθεσία για τα φορολογικά και την ασφάλειας δικαίου και της φορολογικής ασφάλειας, γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα τώρα για τις επιχειρήσεις. Και λέει λοιπόν η Προεδρία της Μάλτας ότι στο μέλλον πρέπει να βελτιωθεί αυτή η ισορροπία. Εσείς πώς το αξιολογείτε το έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μάλλον διορθώνει η ομιλήτρια της Προεδρίας μπορεί να αποδειχθεί και αντιπαραγωγικό για σημεία όπως αναφέρετε εσείς στο CCCTB και πώς θα ε, επιτευχθεί αυτή η ισορροπία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το έγγραφο εμείς δεν το έχουμε. Αλλά μάλλον όταν το πάρουμε θα σας το δώσουμε και εσάς. Κύριε Επίτροπε. Euh, για τον κατάλογο Υπάρχουν πέντε ομάδες εμπειρογνωμόνων οι οποίοι εργάζονται σε αυτό, περίπου 30 άτομα και εξετάζουν 92 δικαιοδοσίες. Θεωρώ και γι' αυτό είπα ότι είμαι ε, έλογα αισιόδοξο για την κατάρτιση του καταλόγου, τα πράγματα πάνε καλά και τα κριτήρια είναι σαφή. Τα κριτήρια αυτά είναι ε, τριπλής φύσεως. BEPS, διαφάνεια και ε, βλαβερές ή στρεβλές φορολογικές πρακτικές. Η πρώτη κατηγορία μπορεί να γίνει αποδεκτή, αν και τα κριτήρια μέσα στο χρόνο θα γίνουν πιο σκληρά σχετικά με το βρώμικο χρήμα κυρία Μύροβα είναι σε καλύτερη θέση από μένα για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής της οδηγίας που προέρχεται από τις υπηρεσίες της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως ο σύνολό της συνειδητοποιεί τις ανησυχίες και τις απορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο όπως είπαμε ανησυχεί ε, έτσι ώστε κάποιες χώρες να μην καλύπτονται. Το συνειδητοποιούμε αυτό και προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο έτσι ώστε να μην υπάρξει αυτή η διάκριση. Μια τρίτη ερώτηση αναφέρθηκε και στα πλαίσια του ανεπισήμου ΕΚΟΦΗΝ στην Μάλτα και το συζήτησα και στη Washington. Η φορολογική δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο και η νομική βεβαιότητα θα έλεγα σε φορολογικό επίπεδο είναι ένα αστείο. Είναι κάτι το βλαβερό ε, γενικά και σε επίπεδο δικαιοσύνης και σε επίπεδο επιχειρηματικότητας, αλλά δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στη νομική σταθερότητα, βεβαιότητα και την καταπολέμηση της διαφάνειας για τη διαφάνεια μάλλον. Το είπα και στη Μάλτα και το επαναλαμβάνω, ο αγώνας μας για την διαφάνεια θα πρέπει να συνοδεύεται και να εξελίσσεται εκ παραλλήλου με τον αγώνα μας για την σταθερότητα. Και όταν βλέπω το CCCTB, ε, βλέπω ακριβώς ότι έχει σαν στόχο και διαρθρωτικά και λειτουργώντας αντίστοιχα για τους υπόλοιπους παράγοντες θα επιτρέψει την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Η σταθερότητα λοιπόν δεν θα πρέπει να είναι άλοθη για την αγνόηση της διαφάνειας. Το είπα και στους Μαλτέζους φίλους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ο Λούντε Κνίτερ Μάια, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Θα κάνω μόνο μία άσκηση, ε, μόνο μία ερώτηση πρώτα απ' όλα να ρωτήσω αν είστε περήφανος για την πρόοδο που έχουμε κάνει. Αν μπορούμε να συγκρίνουμε την πρόοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ. Και το δεύτερο, σε ό,τι αφορά την ε, συμφωνία ΦΑΤΚΑ. Ξέρω ότι η νομική κατάσταση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, γιατί η συμφωνία ΦΑΤΚΑ διαπραγματεύτηκε με τα κράτη-μέλη θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω ποια είναι τα κράτη-μέλη αυτά τα οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, η διαπραγμάτευση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Και η ερώτηση μου λοιπόν τώρα είναι στα... Αφορά την... Α, αφορά τον πραγματικό δικαιούχο και τους δικαιούχους των μετοχών. Το Κοινοβούλιο Α. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η άποψή σας για το θέμα αυτό και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ, πολύ σημαντικό το θέμα και ευχαριστώ και για τη συντομία σας, ο κύριος Επίτροπος. Σας ευχαριστώ για την εκτίμησή σας για τη δουλειά που ήδη έχουμε κάνει, δηλώσατε ότι είστε περήφανος. Πιστεύω ότι είναι σαφές ότι οφείλεται στην καλή μας συνεργασία. Σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία ΦΑΤΚΑ τώρα, θεωρώ ότι ε, εφαρμόζεται το τέλος της α, τραπεζικής μυστικότητας και είναι ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να εξασφαλίσουμε το τραπεζικό απόρριτο, με συγχωρείτε. Όπως εξήγησα προηγουμένως, αυτή η συζήτηση υπάρχει όχι μόνο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκοσμίω. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια έκθεση μέχρι το 2019 σε ό,τι αφορά τη λειτουργικότητα του συστήματος αυτού. Και σε αυτά τα πλαίσια θα αξιολογήσουμε κατά πόσο χρειάζονται επιπλέον μέρη, όπως η επιβολή κυρώσεων ας πούμε, σε περίπτωση μη σεβασμού των ε, υποχρεώσεων αυτών για τα εμπλεκόμενα μέρη. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ε, ρεαλιστικό υπάρχουν συμφωνίες με κράτη-μέλη Είμαστε βεβαίως δεσμευμένοι με αμοιβαιότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα του μόνιμου δικαιούχου, οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές όπως ξέρετε για να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή. Η Επιτροπή έχει προτείνει να μεταρρυθμίσουμε μια τροπολογία στο ζήτημα αυτό, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι φορολογικές αρχές θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και ότι θα υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι με τις πληροφορίες αυτοί συνδεδεμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σε πρόσφατες συζητήσεις συνειδητοποίησαμε ότι η πρόσβαση στους καταλόγους αυτούς που περιέχουν σε όλες αυτές τις πληροφορίες κάποια κράτη μέλη θεώρησαν ότι δεν είναι απαραίτητη. Ίσως θα είναι λοιπόν καλύτερο να προωθήσουμε μια διασυνοριακή πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, στους καταλόγους αυτούς, ούτως ώστε να προωθήσουμε την φορολογική συνεργασία. Υπό αυτές τις συνθήκες θα είναι ίσως δυνατόν να διασαφηνίσουμε συγκεκριμένα στοιχεία, ούτως ώστε να μπορούμε να ταυτοποιούμε το φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από οποιαδήποτε εταιρεία, από οποιαδήποτε φορολογική οντότητα. Και να μπορέσουμε βεβαίως να καταπολεμήσουμε και την νομιμοποίηση χρήματος που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες. Στα πλαίσια αυτά θα περιμένουμε βεβαίως ως ότου το Συμβούλιο να έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις. Προτού να επαναθεωρήσουμε λοιπόν αυτή την, την ενδεχόμενη ανάγκη για επιπλέον προτάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε, κοιτάμε και το ρολόι. Μέχρι 10.30 είχαμε κανονίσει. Αν έχετε λίγα λεπτά παραπάνω, στη συνέχεια συνεδριάζουν οι συντονιστές, να ακούσουμε όλους τους ομιλητές μας. Ο κύριος Μανουέλ Μογέλ, ευχαριστώ κύριε πίτροπε για την παρουσία σας και για το έργο σας, για τη φορολογική δικαιοσύνη. Δύο ερωτήσεις που ήδη τέθησαν, θέλω να κάνω κι εγώ για κάποιες ε, λεπτομέρειες. Η έκθεση αναχώρα έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα της εξίσωσης. Θυμόμαστε τις συζητήσεις και την τελική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έλεγε ότι η φορολογική βάση που έχουμε αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους φορολογικούς παραδείσους της Ευρωπαϊκής Λίστας. Ενώ εμείς στο Κοινοβούλιο αγωνιζόμαστε έτσι ώστε να είναι δημόσια η έκθεση αναχώρα για όλες τις φορολογικές δικαιοδοσίες για να μην είναι πάρα πολύ αδιαφανή και θολά τα πράγματα. Ε, βρέθηκε ένας συμβιβασμός. Ε, για τους φορολογικούς παραδείσους ε, λέτε ότι έχετε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ή μια αισιοδοξία ενώ ταυτόχρονα είστε και σε εγρήγορση. Δεν ξέρω αν συμφωνεί η πολιτική μου ομάδα εγώ πάντω θεωρώ ότι το κριτήριο τη μηδενική φορολόγηση, μηδενικού φορολογικού συντελεστή πλέον δεν θεωρείται ικανό έτσι ώστε να χαρακτηρίζεται μια χώρα φορολογικός παράδεισος. Δεν ξέρω συμφωνείτε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ φιλόδοξη, όπως και το Κοινοβούλιο. Και το Συμβούλιο προσπαθεί να το ξυλώσει λίγο αυτό. Ε, ε, ε ρωτώ λοιπόν. Ε, έκθεση αναχώρα για ε, όλες τις χώρες και τις φορολογικές δικαιοδοσίες. Ε, ε, ξέρω ότι ενδιαφέρεστε πολύ για τη φορολογική δικαιοσύνη και εργάζεστε πολύ προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά το θέμα είναι ότι οι εταιρείε οφείλουν πολύ περισσότερους φόρους ουσιαστικά από εκείνους που καταβάλουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αντίστοιχη οδηγία κατά της φοροδιαφυγής είχε είναι μία ρήτρα switch over, δηλαδή ε, να υπάρχει μια πραγματική φορολόγηση, μια ελάχιστη κατώτατη, να ξέρουμε ποια είναι η φορολογική βάση για ένα ελάχιστο συντελεστή ε, φορολογικό για τη φορολόγηση των εταιριών. Δεν μπορούμε να μιλάμε για φορολογική δικαιοσύνη όταν οι πολυεθνικές στην Ευρώπη πληρώνουν 1% φόρο, για να μην πω λιγότερο. Δηλαδή, κοινή γνώμη πραγματικά αντέδρασε, αλλά και οι βουλευτές. Ε, και ε, μόλις μαθαίνω ότι η Μεγάλη Βρετανία στις διαβουλεύσεις πριν και μετά το Brexit έχει για θέση να εξαιρούνται οι δικές της κτήσεις και τα εδάφη. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Euh. Η Μεγάλη Βρετανία συνεχίζει να παίζει ένα ρόλο επικοδομητικό και σε επίπεδο πρόληψης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Το να δούμε τι είναι ο φορολογικός παράδειγμα. Είναι μια χώρα η οποία δεν σέβεται τα παγκόσμια επίπεδα και τις ρυθμίσεις, ενώ υπάρχουν και χώρες οι οποίες είναι ε, με τον τρόπο τους ανταγωνιστικές στο τομέα των φορολογικών. Εκθέσατε κύριε Μορέλ πολλές ερωτήσεις για την λίστα. Όταν λέγω ότι είμαι επιφυλακτικά αισιόδοξο εμένω σε αυτό. Ε, να διευκρινιστεί καταρχάς η κατάσταση σε σχέση με το μηδενικό επίπεδο επιβολής, ποσοστό επιβολής. Αν τώρα ε, υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζουμε ε, βλαβερό ή βλαπτικό offshoring, αυτό θα φανεί από το screening. Και ταυτόχρονα αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη με το πέρασμα του χρόνου και με τις προόδους που γίνονται για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Κάθε συμβιβαστική λύση έχει τα όρια της, εμείς επιλέξαμε τη συγκεκριμένη γιατί θα επιτρέψει ένα κατάλογο ο οποίος να είναι αξιόπιστο Σχετικά τώρα με, με την έκθεση αναχώρα το δημόσιο κομμάτι. Ε, εγώ ήδη από την πρώτη μέρα της εισόδου μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήμουνα υπέρ της διαφάνειας σε σχέση με τις εκθέσεις αναχώρα και έδωσα μάχη και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταλήξαμε σε μια κριτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι' αυτό. Κάποιοι θεώρησαν ότι οι ρυθμίσεις αυτές ήταν υπερβολικές. Εγώ εμένω στην πίεση και απαιτείται και από πλευρά σας πίεση προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ο να συνεχίζεται, δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις ως προς αυτό. Σχετικά τώρα με, την πραγματική, με το πραγματικό ποσοστό επιβολής όταν μιλάμε για τα CCCTB δεν υπάρχει η ελάχιστη πολιτική βούληση για να επιβληθεί ένα ελάχιστο επίπεδο σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Πρέπει να το διευκρινίσω αυτό. Πολλές χώρες δεν το σκέφτονται καθόλου, δεν θέλουν να το σκέφτονται. Αν θέλουμε να πιέσουμε προς ένα τέτοιο κατώτατο επίπεδο, αυτό θα ήταν αρνητικό για την αναζήτηση μιας συμβιβαστικής λύσης. Θα προτιμούσα τις προτάσεις για ένα ε, πραγματικό επίπεδο επιβολής, έτσι ώστε να μην είναι μηδενική η επιβολή ή ανεπαρκής και από την άλλη η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ορισμένα καθεστώτα φορολογίας τα οποία θεωρούνται επιδοτήσεις κρατικές ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει γιατί δεν θεωρείται κανονικό. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ο Νούνο Μέλο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και έχω κόμμα. Το Ρέμοντ Finch και δύο κατσιάι. Και μετά να κλείσει ο κατάλογος, θα παρακαλούσα. Αν συμφωνείτε κύριε Επίτροπε. Ε, δύο έχω. Ήθελα να κλείσω τον κατάλογο τώρα. Λοιπόν, κύριος Νούνο Μέλο. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ακούσω την ε, θέση σας σε ό,τι αφορά την ε, διαφάνεια για τις διάφορες βάσεις των εταιριών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Λουξεμβούργο, τα Πορτογαλικά νησιά κτλ. Πώς σκοπεύετε να εξετάσετε την ομιμότητά τους ε, και την διαφάνειά τους. Δευτερευόντως, έχουμε ένα διεθνές κέντρο επιχειρήσεων στην Μαδέιρα. Υπάρχει ένα ιδιαίτερα ψηλό χρέος εκεί, 132% του ΑΕΠ της χώρας στην Πορτογαλία. Η το 31% του χρέους θα αποπληρωθεί από Ευρωπαίους φορολογούμενους πολίτες. Και ο χρόνος αποπληρωμής από 15 χρόνια θα ανέβει σε 60 χρόνια. Αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά για τη χώρα μου. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η θέση σας. Ευχαριστώ για τη σύντομη ερώτηση. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε, για τι πορτογαλικέ κρίσεις, ε, ε, Πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό και προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε διαφάνεια παντού σε ό,τι αφορά την φορολογία, σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, την εξέταση καταλόγων σε ό,τι αφορά τους κώδικες διοντολογίας. Υπάρχει μια πρόσβαση πολύ πιο εύκολη, μια μετακίνηση, μια κυκλοφορία δεδομένων, ε, με συγχωρείτε, εγγράφων μεταξύ των διαφορών κρατών μελών. Δεν πρόκειται για μια επανάσταση ό,τι αφορά την διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη ζούμε όλοι μαζί σε μια κοινωνία νέων τεχνολογιών. Όλοι έχουμε στη ε, διάθεσή μας πληροφορίες. Θεωρώ ότι πάντοτε πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Η Επιτροπή, όπως ακριβώς και η δική σας Επιτροπή, εργαζόμαστε από κοινού. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα της Πορτογαλίας, δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για την πορτογαλική πολιτική, δεν μπορώ επομένως να εκφραστώ πάνω στο ζήτημα αυτό. Βρισκόμαστε όμως στη διαδικασία συνεργασίας με την πορτογαλική κυβέρνηση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε το χρέος. Φιλοδοξία μου λοιπόν είναι να επιληθεί το ζήτημα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να μπορέσουμε να μειώσουμε το χρέος, Βεβαίω η Πορτογαλία τηρώντας τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Ένωση. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα του χρέους, είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα. Βλέπουμε ότι οι συζητήσεις πάνω στο ζητούμενο αυτό δεν είναι και πάρα πολύ εύκολες. Καλά, αλλού τις συζητήσεις για το χρέος, όχι εδώ, έχετε δίκιο. Ο Ράιμον Φίντς, τελευταίος, στον κανονικό κατάλογο και μετά τρία κατζιάι. Ένα λεπτό έκαστος. Για να κλείσουμε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την προθυμία σας να παραμείνετε παραπάνω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο αυτό αντιτάσσονται σε σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Τι θεωρείτε για την προοπτική του γεγονότος ότι κάποιες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορεί απλούστατα να αρνηθούν να έχουν ε, ε, να, συνεργάζονται με, με αμερικανικές επιχειρήσεις. Τι πιστεύετε γι' αυτό? Ευχαριστώ πολύ. Δύσκολη ερώτηση αυτή, παρακαλώ. Δεν ξέρω πώς το εννοείτε. Δεν έχω καθόλου την εντύπωση εγώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Κοινοβούλιο να αντιτίθενται στην επιχειρηματικότητα. Εγώ το αντιλαμβάνομαι ως εξή. Εάν το θέμα είναι να θυμίσουμε σε όλους ότι θα πρέπει να φέρονται ε, ως ειλικρινείς και τίμοι φορολογούμενοι και νομοταγείς, και να μην ε, Υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Ορισμένοι είναι υποχρεωμένοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη και οι άλλοι έχουν στρατιέ δικηγόρων, φορολογικών συμβούλων, φοροτεχνικών και είναι σε πλεονεκτική κατάσταση. Προφανώ εκεί ε, θέλουμε να ε, θεσπίσουμε ορισμένου κανόνε που να αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο. Από την άλλη όμω δεν θεωρώ καθόλου ότι ε, πρέπει να φέρουμε αντίπαλες την επένδυση και τη διαφάνεια, την επιχειρηματικότητα και τη διαφάνεια. Χρειαζόμαστε να έχουμε επιχειρήσει να λειτουργούν ε, καλά, εύρωστες, να παραμένουμε ανταγωνιστική οικονομία. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι υπέρ των επιχειρήσεων. Το καλύτερο παράδειγμα ε, είναι η κοινή ενοποιημένη ε, βάση για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, CCCTV. Γιατί ο μηχανισμός αυτός μειώνει το βάρος για τις επιχειρήσεις, απλουστεύει τη ζωή των επιχειρήσεων και διευκολύνει την καταπολέμηση της φοροποφυγής και της φορολογικής απάτης. Πραγματικά σας παρακαλώ, και αυτό είναι ένα πολιτικό μήνυμα από πλευρά μου, ε, υποστηρίξτε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι προς αυτή τη φορολογική βάση θα πρέπει να περάσουμε, που να είναι κοινή αλλά και ενοποιημένη. Επιμένω, στα αγγλικά τρία 3C, δεν είναι δύο, δεν είναι απλώς κοινή βάση, είναι κοινή ενοποιημένη βάση ε, ε, φορολόγηση των επιχειρήσεων. Ακόμα και αν αυτό γίνει σε δύο στάδια, θα πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως η προσπάθεια για τα λοιπά, για τη ΦΑΤΚΑ, η οδηγία DAC 2 θεωρώ που τερματίζει το τραπεζικό απόρριτο είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό. Ο Αμερικανικός νόμος έχει ένα στοιχείο τεροδικίας. Τα κράτη-μέλη δέχτηκαν ε, να τον εφαρμόσουν και σχεδόν όλα έχουν διμερή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι νομίζω ε, πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτό είναι ο σωστός δρόμο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ κύριε πίτροπε Τώρα, από τρία, λεπ... Ε, λεπτά, ένα λεπτό καθομιλητής και αφού απαντήσετε θα ε, λήξει συνεδρίαση. Ένα γκόμες, για ένα λεπτό. Για να επανέλθω στην Πορτογαλία, κύριε Επίτροπε. Η Τρόικα, στην οποία συμμετέχετε, ανησυχεί γιατί ότι εν τω μεταξύ έγινε γνωστό ότι 22 δις ευρώ, το 1 τέταρτο δηλαδή των χρημάτων το οποίο δόθηκε για το πρόγραμμα, πέρασε ε, σε φορολογικούς παραδείσους μέχρι το 2014 χωρίς άλλα φορολογικά έσοδα. Ανησυχεί γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει περισσότερα στοιχεία. Ευχαριστώ και για τις πληροφορίες για το ΦΠΑ. Πράγματι χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία. Θα ήθελα να μου πείτε αν οι ελεύθεροι λιμένες της Σιγκαπούρης, του Λουξεμβούργου και τα λοιπά σας ανησυχούν σαν κέντρα για βρώμικο χρήμα. Ευχαριστώ πολύ, Μπάντ Λούκα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πίτροπε για την ε, φιλική παραδοχή ε, ότι ήταν σημαντικό αυτό που είπα και η συμφωνία μας. Ελπίζω να συμφωνήσουμε και στο μέλλον για τη νομική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άρθρο 125 θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν απαντήσατε ακριβώς στην ερώτησή μου. Για ποιο λόγο τα κράτη-μέλη έχουν τόσους λίγους πόρους που διαθέτουν για να αντιμετωπίσουν τα ύποπτα περιστατικά. Ήσασταν και ο ίδιος υπουργό Οικονομικών στη Γαλλία. Το 1% διεκπεραιώνεται. 400 περιπτώσεις από 40.000. Ε, Βέβαια μπορούν να έρθουν να λένε τα κράτη-μέλη ότι δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή το ποσό που θα εισπράξω ε, από τους φόρους δεν μου καλύπτει όλη αυτή τη διοικητική ε, μηχανή που χρειάζεται να διαθέσω. Μπορείτε να ρωτήσετε στα κρατη Κάπου θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος ε, της απόδοσης και της επιτυχίας. Πόσα φορολογικά έσοδα δηλαδή εισέπραξε το κράτος για το φορολογικό έγκλημα. Και ε, αν το ρωτήσετε αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη, να ξέρουμε ε, πραγματικά τι κόπο κάνουν, τι χρόνο και πόρους αφιερώνουν και τι εισπράττουν. Θα μας βοηθούσε πολύ στη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά και τώρα ο Λουί Μισελ. Και εσείς ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Συγχαρητήρια. Εγώ μπορώ να ε, σας πω γιατί έχω διατελέσει μέλος προηγούμενης επιτροπής. Πρώτη φορά βλέπουμε μια τέτοια ισχυρή θέληση και ισχυρή δέσμευση ε, όπως ε, αυτή που εσείς εδώ επιδεικνύετε. Δύο ερωτήσεις απλές. Πρώτον, έχετε εκτιμήσει καθόλου το ποσοστό των παρανομών κατασκευών σε σχέση με τις νόμιμες μορφές λειτουργίας. γιατί υπάρχουν ε, ορισμένοι τρόποι που μπορεί να είναι ανήθικοι, αλλά είναι ε, νόμιμοι. Δεύτερον, και στο ίδιο πνεύμα, μπορείτε να καταλήξετε σε ένα κοινό ορισμό ε, του τι εστί φορολογική απάτη, φορολογική βελτιστοποίηση, μηχανισμοί επιθετικής φορολογικής πολιτικής και σχεδιασμού. Δηλαδή, όλα αυτά ε, μπορεί να ισχύουν ως ορισμοί, αλλά πολλές φορές ε, τη χάνουν τρομακτικής χειραγώγησης κάποιοι νόμοι. Τελευταίος γύρος ε, απαντήσεων, ο κύριος Επίτροπος, παρακαλώ. Να απαντήσω στην κυρία Γκόμες. Δεν ε, είναι μόνο πορτογαλικό το θέμα σας, αν και προέρχεται από την Πορτογαλία η κυρία Γκόμες. Συμφωνώ με τις ανησυχίες της αυτός είναι και ο στόχος λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής. Τώρα για, τα, για τους ελεύθερους λεγόμενους λιμένες ή λιμένες ελευθέρων συναλλαγών. Free ports. Εγώ είμαι υπεύθυνο και για τα τελωνία και γι' αυτό θα πρέπει η παρακολούθηση αυτών των δραστηριοτήτων να είναι ουσιαστική σχετικά με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Λούκε στα πλαίσια της έκθεσης για τον ΤΑΚ ε, θα συλλέξουμε στατιστικά, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία από όλα τα κράτη-μέλη. Και τα στοιχεία αυτά στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμα αφού τα επεξεργαστούμε. Κάνατε κάποιες εκτιμήσεις τις οποίες θεωρώ απεσιόδοξες. Δεν σημαίνει αυτό ότι θέλω σώνη και καλά να είναι αισιόδοξε. Ίσως να χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις από τα κράτη-μέλη γιατί ο συσχετισμός αυτός είναι πολύ σημαντικός. Για τον κύριο Μισελ με χαρά τον ξαναβρίσκω εδώ και τον ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά του λόγια. Εμείς στην παρούσα φάση δεν έχουμε κάποια εκτίμηση σχετικά με τις ε, νόμιμες και τις μη νόμιμες φορολογικές ρυθμίσεις και προγράμματα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Θα το δούμε και μαζί σας και θα τα δείτε αυτά όταν κάνουμε την πρότασή μας για τους λεγόμενους χρηματοοικονομικούς ενδιαμέσους ή διαμεσολαβητές κτλ. Σχετικά τώρα με τις επιθετικές φορολογικές ευνοϊκές ρυθμίσεις βλέπουμε ποια είναι η διάκριση ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες από τη μία εξαπάτηση της εφορίας. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος δεν σέβεται τις υποχρεώσεις του και δεν εφαρμόζει τον νόμο. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο τον διευκολύνει. Η επιθετική φορολογική, αν θέλετε, πρακτική ή η φορολογική βελτιστοποίηση που είναι συνώνυμη είναι η χρήση υπαρχόντων μηχανισμών νόμιμων έτσι ώστε να επιτραπεί σε επιχειρήσεις, κυρίως πολυεθνικές αλλά όχι μόνο, να ελαχιστοποιήσουν τις καταβολές τους και να πληρώσουν πολύ λιγότερους φόρους, ε, κάτι το οποίο άπτεται και της καταπολέμησης της απάτης, κάθε μορφή δηλαδή διάβρωσης της φορολογικής βάσης, όπως η μεταφορά των κερδών σύμφωνα με τον BEPS Όλα αυτά είναι μία κατηγορία και νομίζω ότι πάνω σε αυτά θα μπορέσουμε να δώσουμε μια πλήρη απάντηση σε εύθετο χρόνο. Εγώ έδωσα μια πολύ γρήγορη απάντηση τώρα, αλλά θα σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία πάνω σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος Επιτροπής μας και για την προθυμία σας να παραμένετε 16 λεπτά παραπάνω από το προγραμματισμένο χρόνο. Έχουμε την αίσθηση ότι στο πρόσωπό σας έχουμε ένα ε, πολύ γερό σύμμαχο για την καταπολέμηση του ξεπλήματος ε, της φοροδιαφυγής, φοροποφυγής. Πολύ θετικό αυτό. Υποστηρίζω και υπογραμμίζω αυτά που είπαν πολλοί συνάδελφοι. Στην αρχή Αναφερθήκατε στην πρόσβαση στα έγγραφα. Αυτό θα το συζητήσουμε τώρα στη συνέχεια στους συντονιστές. Και επίσης είπατε ότι είστε πρόθυμος να ξανάρθετε όταν θα έχετε την πρότασή σας για τους ενδιαμέσους. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο στη δουλειά σας. Πέντε λεπτά διάλειμμα και ακολουθεί η συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών και παρακαλώ να αποχωρήσουν όσοι δεν δικαιούνται να είναι παρόντες στην κυκλισμένη των θυρών συνεδρίες. Ευχαριστώ και πάλι.